Η συζήτηση έληξε. Αύριο 2 Απριλίου θα ξεκινήσουμε στις 9 η ώρα το πρωί και έχουμε δύο συνεδριάσεις. λύεται η συνεδρία. Καλό βράδυ.